Good morning. First point agenda is the... Καλημέρα σας. Πρώτο σημείο η ψηφοφορία για τον ορίζοντα του 2020 και το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με εισηγητή τον κύριο Σοφοκλή Σοφοκλέους. και η Τερέζα Αργέρα Μαντουρέν για την γνωμοδότηση. Σημείο 12, παράγραφος 1, τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος actually. actually. the vote is closed. Έληξε. Εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Πρέπει να αλλάξω γυαλιά. 35. Ψηφίστε ηλεκτρονικός. Όχι, υπέρ, διαχειρός, υπέρ, κατά. Επαλήθευση και πάλι. για να είμαι βέβαιος και για να υπάρχει διαφάνεια γι' αυτό. Ξανά, ποιος είναι υπέρ διανατάσεως, κατά. Ωραία. Θέλω να επαληθεύσω, ρε παιδιά. Ψηφίσατε παρακαλώ. Έληξε. Απαρρίπτεται. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Υπέρ μάλλον. Κατά. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Τριάντα έξι είπαμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεκατέσσερα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά απορρίπτεται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 41 υπέρ κατά απορρίπτεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. και 47 υπέρ κατά απορρίπτεται 48 υπέρ κατά απορρίπτεται 49 υπέρ κατά απορρίπτεται 27 υπέρ κατά εγκρίνεται 50 υπέρ κατά απορρίπτεται 51 υπέρ κατά απορρίπτεται 52 υπέρ κατά απορρίπτεται 28 υπέρ κατά εγκρίνεται 54 υπέρ κατά απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά επαλήθευση για την 56. Έληξε. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ξανά ηλεκτρονικά. Τρεις ακόμη είναι κατά, δεν δουλεύει το μηχάνημα. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. 29 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά εγκρίνεται 61 υπέρ κατά απορρίπτεται 63 υπέρ κατά απορρίπτεται 62 υπέρ κατά εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ένα υπέρ κατά εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά εγκρίνεται. 32 είναι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 31, όχι 7, 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα η τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Έληξε. 32 ψήφοι υπέρ 7 κατά και καμία αποχή. Είχατε ψηφίσει υπέρ και δεν δούλεψε, ναι και εγώ το ίδιο έπαθα. Επόμενη ψηφοφορία. Κανόνες για τον ορίζοντα 2020. Λοιπόν, τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 4 έχει αποσυρθεί, αποσυρθεί. 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά απορρίπτεται. 9 υπέρ. Όχι, έχει αποσυρθεί, έχει αποσυρθεί και η 10. 11 υπέρ. Κατά. Και εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά 33 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Συν τους 4 και εσάς. Εγκρίνεται. Τρίτη ψηφοφορία, η εφαρμογή του προγράμματος Ορίζοντα 2020 τροπολογία 1 γιατί η προηγούμενη είχε αποσυρθεί. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά γκρίνεται 12 υπέρ κατά απορρίπτεται 13 υπέρ κατά επαλήθευση ηλεκτρονικός είναι και οι τέσσερις υπέρ που δεν, έχουν, δεν δουλεύει το μηχάνημά τους. Λοιπόν, λίγη ψηφοφορία. Δεκαεννέα κατά συν τους τέσσερις που δεν δουλεύει το μηχάνημα, 23. Α, όχι, μόνο τρεις, μόνο τρεις. Απορρίπτεται. Δεκατέσσερα υπέρ κατά απορρίπτεται 16 υπέρ κατά απορρίπτεται επαλήθευση α ωραία γιατί όχι περκένω άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται. 19 Δεκαεννέα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Είκοσι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 αποσύρθηκε. 22 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά απορρίπτεται 29 υπέρ κατά απορρίπτεται 30 υπέρ κατά απορρίπτεται Σαράντα ένα υπέρ κατά Απορρίπτεται. Α, όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τρία, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 47 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 48 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά εγκρίνεται εξήντα πέντε Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 68. 69 με 72. Όχι. Α, μία-μία, εντάξει, καλά. 69, υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Έληξε. απορρίπτεται 70 υπέρ κατά επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία έληξε η ψηφοφορία τα ίδια απορρίπτεται 75 υπέρ, όχι 71, 71 υπέρ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Πώς επαλήθευσης Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι και όλες, έληξε η ψηφοφορία. Συν δύο υπέρ. Εγκρίνεται. Όχι καταπίπτει οι φωνές. Μα υπάρχουν άλλοι δύο υπέρ που δεν δουλεύει το μηχανημάτων. των. Από το ΕΛΚ ήταν και οι δύο. Τι ψηφίσατε εσείς κατά και εσείς τρίτη πάλι υπέρ είναι. Φαίνεται δεν έχουμε ξυπνήσει καλά σήμερα. 73. 73 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 74 όμως υπέρ, κατά, εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται τελική και ηλεκτρονική ψηφοφορία. εγκρίνεται πανηγυρικός. Σας ευχαριστώ.